παραλλήλου να δώσω στην κυρία Τζολί τον λόγο. Thank you. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, κύριοι Επίτροποι, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, σας θέτω αυτό το προφορικό ερώτημα σήμερα εκ μέρους της Επιτροπής Ανάπτυξης αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να υποβάλω το ψήφισμα που ομόφωνα εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανάπτυξης. Οι συνάδελφοι της Επιτροπής Ανάπτυξης εργαστήκανε μαζί μου επίπονα για να μπορέσουμε να συζητηθεί αυτό στην Ολομέλεια πριν από το G, τη συνάντηση G20. αλλά Καμία άλλη ομάδα πολιτική δεν υποστήριξε την ένταξη στην ημερήσια διάταξη. Απαραίτητη ήταν η ένταξη αν θέλουμε το Ευρωκοινοβούλιο να παίξει κάποιο ρολό ενισχυμένο στον προσδιορισμό της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχει και δυνατότητα προτάσεων. Αγαπητοί συνάδελφοι, γιατί θα πρέπει να ψηφίσουμε αυτό το ψήφισμα που διατυπώνει τις απόψεις του Ευρωκοινοβουλίου προς την ομάδα των 20 και ειδικότερα προς τα κράτη μας μέλη που συμμετέχουν, καθώς και προς την Κομισιόν. Τι νόημα έχει να ψηφίσουμε μετά το Πίτσπουργκ. Αυτό υπονομεύει το έργο το οποίο έχει πραγματοποιηθεί. Δεν μπορεί να είμαστε απλώ σχολιαστέ τη επικαιρότητα. Δεν είναι αυτό ο ρόλο μα. Α το αφήσουμε αυτό στου επαγγελματίε τους ειδικού, τους δημοσιογράφους δηλαδή. Οι αναπτυσσόμενες χώρες χρειάζονται, μας χρειάζονται τη βοήθειά μας περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση ε, ζημίωσε πολύ σημαντικά τις αναπτυσσόμενες χώρες. Τα περισσότερα δάνεια και πιστώσεις δόθηκαν στην Ευρώπη πολύ λίγες αφρικανικές χώρες μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις για να λάβουν δάνεια. Ε, μόνο 1,6% των δανείων από το ε, Παγκόσμιο Ταμείο ε, μπόρεσαν να εισπράξουν οι αφρικανικές χώρες. Τα υπόλοιπα πήγαν στις ευρωπαϊκές χώρες. Στο διεθνές από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Βεβαίως ήταν πάρα πολύ σημαντικό να ενισχυθούν οι Ευρωπαίοι, αλλά μην ξεχνάμε τη μιζέρια στα σύνορά μας, ε, μιζέρια η οποία ενισχύεται με δικιά μας ευθύνη. Συνεπώ, οι ενισχύσεις για την ανάπτυξη πρέπει να αυξηθούν ταχύτητα, ταχύτατα, τα περισσότερα κράτη από αυτά δεν ανταποκρίνονται στις ε, προϋποθέσεις του ΩΣΑ είναι επίγουσα η κατάσταση και δεν έχουμε χρήματα. Πρέπει να βρούμε δηλαδή νέους πόρους χρηματοδότησης και πηγές χρηματοδότησης, μεταρρυθμίζοντας το σημερινό σύστημα. Η Επιτροπή Ανάπτυξης σας ζητά λοιπόν να ενεργήσετε ώστε να εξαλείψετε τους φορολογικούς παραδείσους, την αποφυγή καταβολής των φόρων και την παροχέτευση των πόρων προς τις βαλκανικές χώρες. Μία νορβηγική έκθεση του Ιουνίου με στοιχεία επαληθευμένα μας λέει ότι τα πιο παράνομα χρήματα που φεύγουν από τις αναπτυσσόμενες χώρες είναι 10 φορές μεγαλύτερα σε ύψος από ότι η ενίσχυση, η αναπτυξιακή που δίνουμε. Συνεπώς, θα πρέπει οι διασυνοριακές επιχειρήσεις να υποχρεωθούν να δηλώσουν τους φόρους που καταβάλουν χώρα, ώστε να έχουμε διαφάνεια του τι καταβάλουν αυτές οι διεθνικές επιχειρήσεις εκεί όπου λειτουργούν. Επίσης πρέπει να μεταρρυθμιστεί το σύστημα με νέες διατάξεις δημοκρατικές και διαφανείς για το εμπόριο και το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα. Οι ευθύνες είναι βαριές. Το πρόβλημα μεγάλο, το έργο δύσκολο, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι ηγέτης στη μεταρρύθμιση αυτών των πράγματων. Ευχαριστώ. Merci. Now the Commissioner De Hucht, please. Ο Επίτροπος De Hucht. Mr. President, uh, dear colleagues. Κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι, η Επιτροπή στο ρόλο της ως εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης του G20 μαζί με την Προεδρία τάσσεται υπέρ της ενισχυμένης ενίσχυσης των ε, χωρών χαμηλού εισοδήματος ως μέλος των δοσμεύσεων του G20 και είναι σημαντικό λοιπόν οι χώρες αυτές να λάβουν επαρκή χρηματοδότηση για να αντιποκριθούν στις ανάγκες που προκύπτουν ιδιαίτερα στα πλαίσια της ε, χρηματοπιστωτικής κρίσης και γι' αυτό Είμαστε υπέρ της βελτίωσης της πρόσβασης από τις ευαίσθητες χώρες χωρίς ε, θεσμικές ε, συχνά ικανότητες και διοικήσεις στις χρηματοδοτήσεις που διαθέτουν διάφοροι διεθνείς οργανισμοί και δωρητές. Εγώ προσωπικά θα ταχθώ υπέρ της ε, μεθόδου αυτής στο Συμβούλιο της Δεκεμβρίου και θα ασχοληθώ ιδιαίτερα με θέματα χρηματοπιστωτικής κρίσης τις επόμενες εβδομάδες. Ελπίζω να έχω την υποστήριξή σας. Στο πλαίσιο αυτό, ο ευαίσθητος χαρακτήρας και τα μέτρα αντιμετώπισης του είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Η Επιτροπή έχει εργαστεί με τον οδικό χάρτη και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για να εντοπιστούν οι πιο αδύναμες χώρες και να συντονιστεί η βοήθεια που παρέχεται από τα δύο αυτά ιδρύματα προκειμένου να περιοριστούν ε, τα προβλήματα. Μεταξύ του 2009 και του 2010 μέχρι 5 δισεκατομμύρια θα δοθούν σε αυτές τις χώρες. Στις χώρες αυτές. Θα ήθελα να σας πω ότι ο μηχανισμός αυτός δεν θα προκαλέσει τέτοια κενά, τέτοια χάσματα, γιατί έχει γίνει σχετική έρευνα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι χώρες που δεν ε, δικαιούνται τέτοια κονδύλια θα προταθούν για άλλα κονδύλια, όπως για παράδειγμα ε, χρηματοδοτήσεις μετά από ad hoc ε, έρευνα των χωρών αυτών κτλ. Σε ό,τι αφορά τον στόχο της ενίσχυσης είμαι βέβαιος ότι η ευελιξία που ήδη υπάρχει επιτρέπει στις παραλεπτρίες χώρες να χρησιμοποιούν τα κονδύλια κατά τον τρόπο που θεωρούν τον πλέον κατάλληλο. Επιπλέον η ενδιάμεση αναθεώρηση θα αποτελέσει μια καλή ευκαιρία να εντοπιστούν οι νέες ανάγκες και να εκτιμηθεί κατά πόσο χρειάζεται περαιτέρω ενίσχυση. Αυτή η ενδιάμεση αναθεώρηση θα δώσει μια επιπλέον ευκαιρία να εξετάσουμε και πάλι τις χώρες ΑΚΕ και κατά πόσο χρειάζονται περαιτέρω ενίσχυση από τα αποθέματα σε ό,τι αφορά την μεταρρύθμιση των Ιδρυμάτων Bretton Woods. Ο ρόλος μας φυσικά είναι περιορισμένος. Το θέμα της εκπροσώπησης θα συζητηθεί στην ετήσια συνάντηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Ταμείου στην Κωνσταντινούπολη, στην οποία θα παρευρεθώ εγώ και ο Επιτροπός Αλμούνια. Επίσης θα συζητηθούν θέματα και υποσαχάριας Αφρικής και θα εξετάσουμε με ενδιαφέρον τις περαιτέρω προτάσεις σε ό,τι αφορά τις παράνομες οικονομικές ροές. Θα ήθελα να πω στην κυρία Ζολή ότι έχω ήδη δώσει εντολές στις υπηρεσίες της Επιτροπής για να ερευνήσουν τέτοιες ροές και να καταπολεμηθούν αυτές οι παράνομες ροές. Και αυτή η κρίση κατέληξε μεταξύ άλλων ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε το μηχανισμό για την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Γιατί αυτό είναι πιο σημαντικό παρά ποτέ. Σε αυτούς τους δύσκολους οικονομικούς καιρούς είναι η ιδιαίτερη ευθύνη που μας βαρύνει ενώπιον του κόσμου προκειμένου η αναπτυξιακή βοήθεια να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά. Στην ανακοίνωση της του Απριλίου η Επιτροπή τόνισε τη σημαντική συμβολή των καινοτομικών μηχανισμών χρηματοδότησης ως μέσα ενίσχυσης σε σχέση με την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Και καταφέραμε να συνδυάσουμε τα μέσα αυτά. Χρησιμοποίησαμε για παράδειγμα ε, μέσα μόχλευσης όπως τα αεροπορικά εισιτήρια θα γίνουν τέτοιες συζητήσεις σε υψηλό επίπεδο μεταξύ άλλων και το Μάιο του 2010 που θα διοργανωθεί από τη Γαλλία και σε αυτά θα εμπλακεί και θα συμμετάσχει η Επιτροπή. Ευχαριστούμε Επίτροπε. Ευχαριστούμε Επίτροπε. Τώρα θα μιλήσουν οι πρόσωποι των πολιτικών ομάδων. Πρώτα απ' όλα ο κύριος Ενρίκη Γκερέρο για τρία λεπτά. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Κοιτάξτε, ε, σήμερα έχουμε την επέτειο ενό έτου ε, από τότε που κατέρευσε η τράπεζα Lehman Brothers Τότε λοιπόν, σύμφωνα με του εμπειρογνώμονε, βρισκόμαστε στα πρόθυρα τη οικονομική κατάρρευση και στα πρόθυρα άλλη ε, σοβαρή κρίση. Η οικονομική κρίση εντατικοποιήθηκε και διευρύνθηκε στην πραγματική οικονομία. Και ζήσαμε ένα χρονικό διάστημα όπου είχαμε αρνητική οικονομική ανάπτυξη και ε, μείωση της απασχόλησης. Αλλά οι αναπτυγμένες χώρες αρχίζουν αυτή τη στιγμή να ξεπερνούν την κρίση. Το έπραξαν, για παράδειγμα, η Γαλλία ή η Γερμανία. Και ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακριβώς σήμερα, ένα χρόνο μετά, παρουσίασε τις οικονομικές της προβλέψεις που δείχνουν ότι στο δεύτερο εξάμεινο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα φύγει από την κρίση και την ύφεση. Όμως, οι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες βρίσκονται ε, στα μέσα της κρίσης και θα εξακολουθούν να βρίσκονται στην κατάσταση αυτή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν, ε, όμως δεν προκάλεσαν την κρίση αυτές οι χώρες. Υφίστανται περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο νόμο τις συνέπειές της. Υφίστανται τις συνέπειες με μικρότερη ανάπτυξη, με περισσότερη ανεργία, με απώλεια θέσεων απασχόληση, με λιγότερε άμεσε επενδύσει, με λιγότερη εξωτερική πίστη, με λιγότερα εμβάσματα από του μετανάστε, με ε, λιγότερη επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια και κυρίω με, περισσότερες, με περισσότερου εμπορικού περιορισμού. Εμεί περάσαμε μία περίοδο όπου ε, η σταθερότητα και η καλή κατάσταση ε, διατηρήθηκε για ένα χρονικό διάστημα αρκετά μεγάλο αλλά αυτές οι χώρες ε, κινδυνεύουν να χάσουν μία δεκαετία ε, αγώνα κατά της φτώχειας. Και αυτό σημαίνει μια ολόκληρη γενιά. Μπορούμε να κάνουμε πολλά για να βοηθήσουμε τις χώρες αυτές ε, σε πολλούς τομείς. Και εγώ θα ήθελα να αναφέρω ιδιαίτερα την αντιμετώπιση του προστατευτισμού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την περασμένη εβδομάδα παρουσίασε την τέταρτη έκθεση για τα περιοριστικά μέτρα στο εμπόριο. Εκεί αποδεικνύεται ότι πολλές χώρες υιοθετούν νέα προστατευτικά και περιοριστικά μέτρα. Και αυτό έχει καταστροφικές συνέπειες για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Επίσης, πολλές αναπτυγμένε χώρες δεν ε, ε, ε, εκπληρώνουν τις επίσημες δεσμεύσεις τους για την επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια. Ακριβώς σήμερα που χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ νέους πόρους για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης. Γι' αυτό ε, προτείνω να αυξήσουμε τον ε, συντονισμό της αναπτυξιακής βοήθειας με μια πιο διευρυμένη συμφωνία ανάμεσα στους, στις χώρες που είναι δωρητές, ε, στους, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και στους εταίρους με περισσότερη διαφάνεια έτσι ώστε ε, ε, ε, Χωρί όμω κόστο και, χωρίς, και με λιγότερη γραφειοκρατία. Απευθύνω έκκληση σε όλους και στον Επίτροπο να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση του, του, μέσου που μας παρουσιάσατε και πιστεύω ότι θα συμφωνήσει και ο επίτροπο κύριο Σαλμούνια. Σας ευχαριστώ. Ο Λου, κύριος Λουί Μισελ έχει το λόγο. Για τρία μισή λεπτά. Κύριε Επίτροπε, Κυρία Πρόεδρε της Επιτροπής Ανάπτυξης, βεβαίως έχω συνείδηση του γεγονότος του σε ένα τέτοιο τύπο συζήτησης. Ε, έχουμε επαναλήψεις πολλές. Αυτό όμως δεν με ενοχλεί. Είναι σημαντικό να επαναλαμβάνουμε αυτή την έντονη συνένεση που χρειάζεται το Ευρωκοινοβούλιο να δημιουργήσει με την Κομπισιόν. Ε, ειδικότερα δε σε σχέση με αυτή τη χρηματοπιστωτική κρίση. Υποτίθεται ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες δεν θα θυγόντουσαν από την κρίση. Σήμερα όμως το αποτέλεσμα είναι το αντίθετο. Οι εμπειρογνώμονες λένε ότι θα είναι καταστροφικά τα αποτελέσματα της κρίσης και όλες οι φτωχότερες ε, οι φτωχότεροι πληθυσμοί θα έχουν πτώση της ανάπτυξης και επιδείνωση της φτώχειας. Κύριε Επίτροπε, Χαίρομαι που αναφερθήκατε στην ανάγκη να ανταποκριθούμε κατά τρόπο, τρόπο πιο εύκομπτο σε αυτές τις ανάγκες. Όπως ίσως ξέρετε, πάντοτε προασπιζόμουνα, όποτε ήταν εφικτό με έλεγχο βέβαια, ήμουνα πάντοτε υπερασπιστής της άμεσης ενίσχυσης, της κλαδικής ενίσχυσης, της δημοσιονομικής ενίσχυσης. Ε, υπάρχει ένα αποτέλεσμα πιο θετικό με αυτόν τον τρόπο. Είναι κατάλληλα μέσα στα κράτη. Το, η ομάδα των 20 όμως δεν μεταρρύθμισε τους χρηματοπιστωτικούς μηχανισμούς ε, το Διεθνές Νομισματικό Τομείο, την Παγκόσμια Τράπεζα για να λάβει υπόψη τους ε, τα αποτελέσματα το 80 και τόσο των πρόσφετων δανείων πήγανε στις ευρωπαϊκές χώρες και μόνο 1,6% των δανείων πήγε σε αφρικανικές χώρες. Τα μέσα που υποσχεθήκανε στην ομάδα των 20 για την Αφρική δεν θα επαρκέσουν, το ξέρουμε και δεν θα απευθυνθούν στις πιο στις ασθενέστερες χώρες και δεν θα φτάσουν και εκεί γρήγορα. Η πραγματική πρόκληση, κύριε Πίτροπε, είναι και το ξέρετε, να επιμείνουμε τα κράτη-μέλη να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους του 2005. Δεν μπορούμε να μειώσουμε την κρατική ενίσχυση για την ανάπτυξη. Πολλά κράτη-μέλη όμως ε, ανακοίνωσαν μειώσεις. Η Ιρλανδία 10%, η Ιταλία μείωση 50%, η Λετωνία μείωση 100%. Αυτή τοποθέτηση να απαράδεκτη και ανεύθυνη. Θα ήθελα την άποψή σας λοιπόν για διάφορα ζητήματα. Άκουσα τη θετική σας ε, ανταπόκριση στο, για το Ταμείο ε, που θέλει να δημιουργήσει η Παγκόσμια Τράπεζα για τους ευάλωτους. Επίσης μιλήσατε για τους φορολογικούς παραδείσους. Ε, χώρες χάνουν δισεκατομμύρια ευρώ που μεταφέρονται σε, σε φορολογικούς παραδείσους. Μιλήσαμε για τη διακυβέρνηση, αλλά υπάρχει ακόμη ένα ερώτημα που πρέπει να υπογραμμίσουμε, το εξή: Η ενίσχυση προς το εμπόριο. Εγώ είμαι θερμός υποστηρικτής των συμφωνιών συνεργασίας αρκεί να λαμβάνουμε υπόψη μας τις συγκεκριμένες ανάγκες, αρκεί να υπάρχουν μεταβατικές περίοδοι και αρκεί ε, να τηρούν την υπόσχεσή τους για ένα δις χρόνο όπως υποσχέθηκαν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το εμπόριο κάθε χρόνο. Πολλές χώρες λένε έχουν, ε, λένε πολλά καλά πράγματα για τις αναπτυσσόμενες χώρες αλλά τίποτα δεν κάνουν από την άλλη πλευρά. Με κινησμό μειώνουν τις ενισχύσεις. Ευχαριστώ. Γκάμπι Τσίμερ από την ΚΟΕ. 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Για την προφορική ερώτηση της κυρίας Ζολή μας φέρνει στο σημείο αυτό το οποίο μας απασχολεί ως ε, πολιτικούς. Οι υποσχέσεις των τελευταίων συναντήσεων G8 και G20 τελικά έμειναν ε, στη θεωρία. Ποτέ δεν ε, έχουν οδηγήσει σε επαρκή βοήθεια. Υπό την έννοια αυτή δεν μπορώ να καταλάβω λοιπόν γιατί το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν μπορεί να τύχει διαπραγμάτευσης πριν από το Πίτσμπουργκ ε, για να υπάρξει επιτέλους επαρκής πολιτική πίεση. Νομίζω ότι έγιναν σωστές αναλύσεις και από την Επιτροπή και από τον Λουίς Μισελ. Μου φαίνεται λοιπόν ότι με σαφήνεια προκύπτει ότι ξέρουμε τι φταίει, αλλά δεν είμαστε σε θέση πολιτικός πώς να ασκήσουμε πίεση στα κράτη-μέλη προκειμένου να γίνει μια μεταστροφή και να προωθήσουμε την πολιτική αυτή. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα μεγάλο κίνδυνο εν ώψη του Πίτσμπουργκ. Αν δεν καταφέρουμε να επιβάλλουμε μεγαλύτερη πίεση για το ότι χρειαζόμαστε καινούργια ιδρύματα προκειμένου να στηρίξουμε τι πλέον φτωχέ χώρε, πάλι εδώ θα έρθουμε μετά το Πίτσμπουργκ και θα διαπιστώσουμε ότι δεν έχει κινηθεί τίποτα. Δεν έχει σημειωθεί καμία πρόοδο. Γι' αυτό λοιπόν σα παρακαλώ, Επίτροπε, άμεσα να τοποθετηθείτε εδώ στο Κοινοβούλιο αναφορικά με τα αποτελέσματα και να μας πείτε τι μπορούσαν να πετύχουν τα κράτη-μέλη και τι πετύχαμε. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι γρήγορη και αποτελεσματική δράση. Γιατί μπροστά στα μάτια μας πεθαίνουν άνθρωποι. Και είμαστε εν μέρη και εμείς υπεύθυνοι. Γι' αυτό λοιπόν σας ε, καλώ να δράσουμε από κοινού. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Κυρία Κρέτου. Ευχαριστώ. Ε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Ε, 4,8 δις παρουσιάζει μείωση ε, η, ε, η παροχή βοήθειας προς τις χώρες αυτές. Κοιτάξτε, έχουμε μεγάλη διαφορά ανάμεσα στα κονδύλια τα οποία απαιτούνται και στα κονδύλια τα οποία προέρχονται από τους δωρετές. Από τους δωρετές και ταυτόχρονα δεν μπορούμε ε, παρά ε, να, μην, ε, ε, να μην λάβουμε υπόψη το γεγονό αυτό για να καταλάβουμε πόσα χρήματα δαπανώνται σε άλλου τομεί. πραγματικά κάθε χώρα έχει τα προβλήματά τη, αλλά δεν, είναι, δεν μπορούμε, είναι απάνθρωπο να μην σκεφτόμαστε και τι ε, χώρε αυτέ που αντιμετωπίζουν τρομερή κρίση για την οποία δεν ευθύνονται, ευθύνονται σε λιγότερο βαθμό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ε, ιδιαίτερα κατά την περίοδο της ύφεση ε, ε, θα μειωθεί ακόμα περισσότερο η ανθρωπιστική βοήθεια. Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό, γιατί διαφορετικά η αναπτυσσόμενη φτώχεια θα έχει αποτέλεσμα boomerang και θα έχουμε τεράστιες, τεράστια μεταναστευτικά ρεύματα προς τις αναπτυγμένες χώρες. Λαμβάνοντας υπόψη όλα αυτά, πιστεύω ότι απαιτούνται σημαντικές προσπάθειες προς την κατεύθυνση αντιμετώπισης των ευθύνων ευθυνών μας και της ε, προώθησης ε, της κινητοποίησης της διεθνούς βοήθειας. Ταυτόχρονα θα πρέπει να μειωθεί η εξάρτηση ε, της ανθρωπιστικής βοήθειας από ορισμένε προϋποθέσεις και, τελείως, και τέλος θα πρέπει να ληφθούν υπόψη αυτά τα οποία είπε και ο κύριος Λουί Μισελ, ο πρώην Επίτροπος, για την ανάγκη μεγαλύτερης συμμετοχής της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ε, και ρωτώ, ε, θα προταθεί κάτι στη Σύνοδο Κορυφή ε, αυτή τη Κωνσταντινούπολη. Και θέλω τελειώνοντα να εκφράσω τι ευχαριστίε μου Ε, για αυτά τα οποία είπατε, για τις διάφορες επισκέψεις που έχετε προγραμματίσει για την Αφρική, για το Ζιμπάμπουε, για την επίγουσα βοήθεια ε, για τα 100.000 ε, θύματα της πλημμύρας στην Δυτική Αφρική. Αλλά να σας πω και τέλος ότι όχι μόνο η Μπουρκίνα Φάσο αντιμετωπίζει φυσικές καταστροφές, αλλά και ο Νίγηρας. Και εδώ απαιτείται διεθνής συνδρομή. Και όχι μόνο οι πλημμύρες απειλούν τις ζωές των ανθρώπων, αλλά οι πυρκαγιές, και ε, χαίρομαι για αυτά τα 53 εκατομμύρια που δώσατε την περασμένη εβδομάδα για τις υποσαχάριες χώρες και, υποσαχάριες χώρες και την αντιμετώπιση της ξηρασίας. Ελπίζω λοιπόν όλα αυτά τα οποία ε, ήδη έχετε ξεκινήσει ε, να μεταφερθούν και στη συνδιάσκεψη της Κοπεχάγης και στο Πίτσμπουργκ γιατί αυτές οι συναντήσεις είναι κρίσιμη σημασία. Σας ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστώ και τώρα ε, περνάμε στις παρεμβάσεις του ενός λεπτού. Η κυρία Ρόιτοβα θέλει το λόγο. Για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ. Ε, κύριε Πίτροπε, θα ήθελα να εκφράσω την απογοήτευσή μου γιατί οι υποσχέσεις ε, τη ε, ε, G20 για βοήθεια προς τις χώρες αυτές χαρακτηρίζονται από έλλειψη σοβαρότητα. Διότι μέχρι στιγμή η βοήθεια είναι απειροελάχιστη. Ταυτόχρονα απευθύνω έκκληση έτσι ώστε να μεταρρυθμιστεί το σύστημα, το σύστημα λήψης αποφάσεων για, και, να, να μεταρρυθμιστεί και το, και το σύστημα Bretton Woods. Τέλο ρωτώ το εξή κυρίω στο, στο, στο επίπεδο τη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και τη παιδεία. Ε, εδώ απαιτείται ιδιαίτερη προσπάθεια για να μπορέσουν οι χώρε αυτέ να αντιμετωπίσουν την κρίση. Ε, είναι δραστική η μείωση τη βοήθεια από τι ευρωπαϊκέ χώρε και αυτό είναι ιδιαίτερα λυπηρό. λυπηρό. Πέραν τούτου, σα εύχομαι κάθε επιτυχία στα καθήκοντά σα. Σα ευχαριστώ γιατί ε, τηρήσατε το ένα λεπτό. Και τώρα... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό και το συζητάμε σε μια σημαντική χρονική στιγμή. Όχι μόνο επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει σαφή αντίληψη του τι θέλει να κάνει με την αναπτυξιακή βοήθεια, αλλά επειδή ακόμη πρέπει να επεξηγήσουμε το ζήτημα και στους λαούς μας. Η αναπτυξιακή βοήθεια και η χρηματοδότησή της μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τη μετανάστευση, τις επιδημίες, τους λοιμούς και όλα αυτά τα έχει εξηγήσει βέβαια το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ε, αλλά τα σωστά προσανατελισμένα χρήματα θα είναι υποφελή για όλους και για τους δωρητές και για τους λαμβάνοντες. Ζούμε σε ευρωπαϊκές χώρες, ακούμε αρνητικά σχόλια βεβαίως για την αναπτυξιακή μας βοήθεια και όσον αφορά τη χρήση αυτής της βοήθειας δεν υπάρχει απόλυτη συνένεση μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών. Θα πρέπει να βρούμε τρόπο να προσανατολίσουμε. Τέλος, η κυρία Καφάια, που είναι πάρα πολύ δραστήρια απόψε βλέπω. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτό το στάδιο η Ευρώπη να δείξει ότι μπορεί να αναλάβει το ρόλο του υπεύθυνου ηγέτη και θα πρέπει ταυτόχρονα να φροντίσουμε έτσι ώστε να τηρηθούν όλε οι δεσμεύσει που έχουν αναλυφθεί και οι στόχοι τη χιλιετία. Είδαμε το πώ ε, οι περισσότερε φτωχέ χώρε ε, πλήττονται ιδιαίτερα σε περιόδου κρίση και ε, κυρίω σε επίπεδο απόλυτη στόχη, εκεί όπου οι άνθρωποι πεθαίνουν από την πείνα και από τι ασθένειε. Κοιτάξτε, ε, ε, ήδη αρκετέ χώρε εξέφρασαν τη βούλησή του ε, για μείωση της ενίσχυση, τη βοήθειας. Μα τώρα επίκει περισσότερο από ποτέ να υπενθυμίσουμε την ανάγκη να υπάρξει καλύτερο συντονισμός και βέλτιστη αξιοποίηση των χρημάτων αυτών. Για παράδειγμα, ένα πρόγραμμα πληροφοριακό το οποίο εφαρμόστηκε στη Μοζαμβίκη ε, ε, πρόγραμμα πληροφορική, συγγνώμη. Μπορούμε λοιπόν ε, και με λιγότερα μέσα, όταν βλέπουμε να μειώνονται οι συνθήκε, να αξιοποιήσουμε αποτελεσματικά τα χρήματα αυτά. Σα ευχαριστώ και τώρα να δώσω το λόγο στον Επίτροπο. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, συνάδελφοι. Ναι, η κρίση έχει χτυπήσει τις πλέον φτωχές χώρες με τον πιο σκληρό τρόπο πιο πολύ από τις άλλες και όντως δεν μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά. Μπορούμε να συζητήσουμε μόνο ποιε είναι οι καλύτερε λύσει να την αντιμετωπίσουμε και προφανώ αυτό θα πάρει πιο πολύ χρόνο από ό,τι θα πάρει στον αναπτυσσόμενο κόσμο γιατί οι μηχανισμοί παραγωγής οικονομικού κέρδους είναι πολύ πιο αναπτυγμένοι. Ένα από τα σχόλια που έκαναν διάφορα μέλη του Κοινοβουλίου είναι ότι πολλά κράτη-μέλη κάνουν πίσω, υπαναχωρούν σε σχέση με τις ε, δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει για την επίσημη μεταξυβική βοήθεια. Τα κράτη-μέλη συμφώνησαν το 2005 0,51% για την Ευρώπη το 15 και 0,7% για την Ευρώπη των 12, για τα νέα κράτη-μέλη. Αυτό ήταν ο στόχος μέχρι το 2010 και 0,7% και 0,33% μέχρι το 2015. Οι χώρες που είχαν ήδη πετύχει υψηλότερα επίπεδα δεσμεύτηκαν να τα διατηρήσουν. προκειμένου από κοινού τα κράτη-μέλη μέχρι το 2010 να έχουν φτάσει σε επίπεδο 0,56% επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας μέχρι το 2010. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την κρίση ως δικαιολογία για να επαναχωρήσουμε και θα παραμείνουμε δεσμευμένοι για να διατηρήσουμε τα επίπεδα που έχουμε υποσχεθεί σε ό,τι αφορά την βοήθεια. Το 2008 αυξήθηκε κατά 4 δισεκατομμύρια σε επίπεδο 0,4% και αυτή η αυξητική τάση προβλέπεται να συνεχιστεί. Βάσει των στοιχείων που έχουμε, προβλέπεται αύξηση σε 53,4 δισεκατομμύρια το 2009, 0,44% και 58,7 δισεκατομμύρια, 0,45% του 2010. Αυτό σημαίνει ότι χωρίς επιπρόσθετα μέτρα από τα κράτη-μέλη για τους μεμονωμένους στόχους, ο συλλογικός στόχος για το 2010 δεν θα επιτευχθεί. Οι προβλέψεις για την αύξηση της ε, αναπτυξιακής βοήθειας εξαρτάται από τις χώρες που καταβάλουν προσπάθειες. Χρειάζονται προσπάθειες από όλα τα κράτη-μέλη όμως και θα συνεχίσω να επιμένω σε αυτό το σημείο γιατί είναι η ευθύνη των κρατών μελών αυτών και είναι μια δέσμευση που έχουν αναλάβει. Και η κρίση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογία για να αποδυναμώσει τις δεσμεύσεις που έχουν λάβει. Πολλά μέλη τόνισαν την ανάγκη ε, μεταρρύθμισης των ε, πιστοτικών ε, ιδρυμάτων. Uh, Αυτό είναι ο στόχος που μπορούμε, με τον οποίο μπορούμε να είμαστε απόλυτα σύμφωνοι. Ε, EG20 ε, καθορίσει, έχει καθορίσει ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ε, για ε, μεταρρύθμιση της διακυβέρνησης και του συστήματος Bretton Woods ζητώντας να επιταχυνθούν και τα σχέδια για τη μεταρρύθμιση πριν δηλαδή από τη Σύνοδο Κορυφής του Λονδίνου. Αναμένονται ορισμένα αποτελέσματα μέχρι τον Απρίλιο του επόμενου έτους από τον Απρίλιο του επόμενου έτους και εγώ πιστεύω ότι θα βρεθούν λύσεις στα εκρεμή ζητήματα. Δεδομένης ε, της ε, υφιστάμενης κρίσης, ε, ε, και ε, της συνδιάσκεψης των G20, η Επιτροπή τονίζει το, τη, την δεύτερη φάση μεταρρυθμίσεων της Παγκόσμιας Τράπεζας, έτσι ώστε να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2010. η Σύνοδος Κορυφής του Λονδίνου στις 2 Απριλίου του 2009 θα μείνει στην ιστορία ε, μια διάσκεψη όπου αντιμετωπίστηκαν τα ζητήματα ανάπτυξης ε, και η παρουσία, ε, όπου και όπου υπήρξε παρουσία εκπροσώπων των υψωμένων χωρών. Προετοιμάζοντα την επόμενη σύνοδο των G20, οι τελευταίοι αυτοί μήνες χαρακτηρίστηκαν από ιδιαίτερη δραστηριότητα ε, και τον Αύγουστο το το, ε, ε, το Διοικητικό Συμβούλιο ε, του Παγκόσμιου Νομισματικού Ταμείου ενέκρινε περαιτέρω 250 δις, από τα οποία 18 δις θα πάνε στις ανεψόμενες χώρες, στις χώρες με πολύ χαμηλά εισοδήματα και όλα αυτά αποτελούν ιδιαίτερα θετικές εξελίξεις. Ο κύριος Λουί Μισελ, ο προκάτοχός μου, τόνισε ιδιαίτερα το θέμα της ευελιξίας, λέγοντας ότι οι, μηχανι... οι δημοσιονομικοί μηχανισμοί στήριξη ε, είναι ε, το πιο ευέλικτο μέσο το οποίο έχουμε. Ναι, ενδεχομένω αυτό είναι αλήθεια. Αλλά αυτό ταυτόχρονα σημαίνει ότι πρέπει να αντισταθμίσουμε Μάλλον θα πρέπει με τους ομολόγους μας στις ανεψόμενες χώρες να ε, δούμε το πώς θα εγκαθιδρύσουμε και θα θεσπίσουμε ένα πολιτικό διάλογο και το πώς θα εφαρμόσουμε και μηχανισμούς παρακολούθησης. Όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι συνεπάγονται ε, μία, ένα ελάχιστο βαθμό συνεργασία και από τις χώρες αυτές. Πάντως και εγώ πιστεύω ότι Ιδιαίτερα ο τομιακό δημοσιονομικό μηχανισμό στήριξη είναι μια άκρο αποτελεσματική διαδικασία. Τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω πολύ καλά γιατί αυτό το ψήφισμα ε, που συζήτησε η Επιτροπή Ανάπτυξης και που αναφέρεται στη συνεδρίαση ε, στο Πίτσμπουργκ δεν ενεκρίθη πριν από τη συνεδρίαση των G20 στο Πίτσμπουργκ. Ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έγινε κάτι τέτοιο. Μάλλον κάποια τεχνική φύσεω εξήγηση θα υπάρχει. Πάντω, κατά την άποψή μου, δίνεται το λανθασμένο μήνυμα από το ε, νεοεκλεχθέν ε, κοινοβούλιο. Ότι δηλαδή θα συζητήσει ένα τόσο σημαντικό ψήφισμα μετά από την σύνοδο στο Πίτσμπουργκ αν δεν κάνω λάθο θα γίνει ε, ε, στο διάστημα 22 με 24 Σεπτεμβρίου. Άρα, πριν την επόμενη Ολομέλη στο Στρασβούργο του Οκτωβρίου. Βεβαίω δεν είναι δική μου αρμοδιότητα, αλλά πρέπει να σα πω ότι και εγώ, όπω και οι άλλοι συναδελφοί σα που εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά του για αυτήν την κατάσταση, πιστεύω ότι είναι κρίμα που δεν μπορέσατε στη συμμετείνα σε αυτή τη σύνοδο να ψηφίσετε το ψήφισμα. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Επίτροπε. Θα ήθελα να αναφέρω ότι η απόφαση αυτή λήφθη από τη διάσκεψη των Προέδρων για την ε, ψηφοφορία τον Οκτώβριο δηλαδή. Γιατί τον Οκτώβριο θα γίνει και συζήτηση και για το G20. Αυτό ως επεξήγηση για την ερώτησή σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συζήτηση αυτή. Λίγη για το θέμα αυτό, όπως ανέφερα.